А, gal pradėsim, ja? Maybe we'll start, Yes, we can start. Uh, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, λοιπόν. Θα μιλήσω λιθουανικά. συνεχίζει λιθουανικά η Πρόεδρος, πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, δύο αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Για το σημείο 6 διαγράφεται γιατί δυστυχώς ο Γαλ, η Γαλλίδη υπουργό, η Λορένσο Ροσινιόλο, δεν θα μπορέσει να έρθει. Και το σημείο 10 διαγράφεται από την ημερήσια διάταξη Πρόκειται για σύσταση της Επιτροπής για τη θέση των γυναικών. Ε, πρόκειται για ψηφοφορία, αλλά θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Συμφωνείτε με τις τροποποίησεις αυτές? Καλώς. Οπότε περνάμε στο σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεων της 9ης Ιανουαρίου 2017. Σημείο 4. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Μία ανακοίνωση έχω. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή μας εφ' θα εφαρμόσει την αρχή paperless, χωρίς χαρτιά. Δηλαδή η ψηφοφορία και όλα τα άλλα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στο ίντερνετ και στο ίντερνετ, αλλά όχι σε χαρτί. Δεν θα έχετε αντίγραφα δηλαδή στην αίθουσα. Μόνο το σχέδιο εμερήσιας διάταξης θα είναι διαθέσιμο σε χαρτί. Και συνεχίζουμε και περνάμε στην ψηφοφορία. Είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε όλοι. Έχετε την κάρτα ψηφοφορίας. Αρχίζουμε. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγητής Ερνέστ Ούρτεσιν. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία, θα ελέγξουμε. Συμβαστική 26. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Διανατάσεως της χειρός τώρα. Τροπολογία 181 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 175 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 166 υπέρ, κατά, Η 166 είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 187 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία. Διακόπτη πρόεδρος. Δεν ε, δούλεψε το μηχάνημα, αυτό ήτανε. Τι ψηφίσατε, υπέρ ή κατά. Υπέρ. Καλώς. 187 ήταν, ναι. Εγκρίθηκε. 16-10 το αποτέλεσμα. 188 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 195 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίφθηκε. 196 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 200 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 209 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 234 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, 45 διορθώνει πρόεδρος, 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 246 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 249 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 48α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σαράντα εννέα συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 270 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 275 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 38 πρώτα. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 με προφορική τροποποίηση. Ναι, Αποσύρθηκε 73 η τροπολογία, οπότε χωρίς αυτή την ε, τροπολογία, χωρίς εκείνη που λέει ότι θα, η εγγύηση θα παίξει ρόλο σε όλες Αυτό βγαίνει από το συμβασμό, γιατί αποσύρθηκε της κι αλλιώς η προφορική. Συμβαστική 11 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 και 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 120. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 και 123 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 133 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 και 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 και 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 20 και 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 24, 25 και 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ,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 Πέρας της φοφορίας, Α, οι σοσιαλιστές ψηφίζουν παραπάνω, παραπάνω όπως θα έπρεπε. Δύο παραπάνω ψηφίζουνε. Τώρα είναι εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Μπράβο, εγκρίθηκε, συγχαρητήρια.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 Η επόμενη έκθεση αφορά την ε, οδηγία του Συμβουλίου σε σχέση με την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Η Αγνιέσκα Κοσλόφσκα Ραγεύιτς είναι η συγγήτρια. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 2 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, βεβαίως ελέγχουμε. Τραν 2 ελέγχουμε. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε έναν σοσιαλιστή, έναν υπεράριθμο. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 71 και 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Με συγχωρείτε. 31. Τραν 31. Υπέρ. Α, δεν ψηφίζουμε, δεν την ψηφίζουμε, όχι, την Τραν 31. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τραν 29. Θέλετε να ελέγξουμε. Τραν 27 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας σοσιαλιστής υπεράριθμος, ο συνήθως, ο συνήθως, σε αυτή την επιτροπή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τραν 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε τραν 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 87. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ με συγχωρείτε, 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 98, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 99 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία για την 104. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία, ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 116 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 5 και 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Θέλετε να ελέγξουμε τις δύο τροπολογίες. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνονται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, εγκρίνεται συγχαρητήρια. σε ό,τι αφορά τι ε, ε, συνθήκες απασχόληση, ε, ο κύριο Ζωάπη είναι ο εισηγητή. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά απόχε. Παρακαλώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 54. «54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε». 58. Σε τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 72. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. 81 ένα υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 συγγνώμη για την 94 να ψηφίσουμε το δεύτερο κομμάτι της, ε, το δεύτερο τμήμα της 94 μα ένα τμήμα βλέπουμε μόνο η 96 έχει δύο τμήματα Okay. Okay, okay, okay. Amendment 96. 96. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Η 2. Υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, να, να ψηφίσουμε το σύνολο του σχεδίου. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας ε, στην συνεδρίαση αυτή και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας και μην ξεχνάτε ότι στις 28 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρία.